Dear colleagues, we... Συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Τώρα το απόγευμα θα συζητήσουμε το πακέτο για την κυκλική οικονομία. Έχουμε πολλά σημεία στην ημερήσια διάταξη από το 8 στο 11. Προτείνω να τα συζητήσουμε όλα μαζί. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από την τροποποίηση δίνοντας το λόγο στον συγκητή, για να μας δώσει σαφή εικόνα για τις τροπολογίες. Η κυρία Μποναφέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την υποβολή τροπολογιών. Αρκετές υπευλήθησαν, 1.700 περίπου για τις τέσσερις οδηγίες. 1.100 μόνο, 1.169 για μία οδηγία, για την οδηγία πλαίσιο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους αυτό δείχνει ιδιαίτερη προσοχή για το θέμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό ζήτημα και η υποβολή τόσων τροπολογιών είναι μάρτυρας του ενδιαφέροντος. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που εργάζονται συνεδριάσεις των σκιωδών, όλους τους σκιώδης ηγητές. Τους ευχαριστώ για ένα κλίμα πολύ ε, συνεργατικό και επικοδομητικό. Ελπίζω να συνεχιστεί και στη συνέχεια των εργασιών μας που θα είναι εντατικής μορφής και μακρά διαρκείας. Στόχος μια θέση με τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε ισχυρή εντολή για συζητήσεις με το Συμβούλιο, διότι από τις φήμες των τελευταίων εβδομάδων φαίνεται το Συμβούλιο καταλήγει σε κάποιες θέσεις που θέλουν να δώσουν νέα διάσταση στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίω από τι χώρε που πηγαίνουν καλά, κυρίω τα βέστα θέματα, όπω είναι οι στόχοι, η μεθοδολογία υπολογισμού και οι ελάχιστε απαιτήσει όσον αφορά την εκτεταμένη ευθύνη του παραγωγού. Πάμε στην ουσία τώρα των τροπολογιών. Είμαι πολύ ικανοποιημένη και από αυτή την άποψη. Οι συνάδελφοι σε μεγάλο βαθμό συμπεριέλαβαν το πνεύμα της εκθέσεώς μου και σε κάποιες περιπτώσεις οι προτάσεις μου ενισχύθηκαν. Ήταν θετικό το αποτέλεσμα. Όσον αφορά δύο στόχους, όλος ιδιαίτερος ε, κεντρικούς κατά την απόψή μου για το πακέτο της κυκλικής οικονομίας. Πρώτα απ' όλα θέλουμε ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και δεύτερον την αγορά των πρώτων υλών και των δευτερογενών υλών. Τώρα για τα μέτρα πρόληψης. Η πρόληψη είναι το πρώτο βήμα στην ιεραρχία αυτή των αποβλήτων και θέλω να πω ότι κανένας δεν αφισβήτησε την ιεραρχία των αποβλήτων που είναι κάτι που ισχύει. Η πρόληψη είναι το πρώτο βήμα. Ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η πρόληψη Όσον αφορά την πρόληψη, η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την άποψή μου, αλλά και κατά την άποψη των συναδέλφων, ήταν κάπω ελλειπή. Και οι τροπολογίε που υπευλήθησαν την ενισχύουν. Όπω προέβλεπα και στην έκθεσή μου, πολλέ τροπολογίε ζητούν από τα κράτη-μέλη προσπάθειε για να ευνοήσουν την παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων που είναι πιο αποδοτικά από πλευράς χρήσεως πόρων δηλαδή προϊόντα ανακυκλώσιμα, επισκευάσιμα ε, που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Και έχουμε άλλα δύο σημεία για την πρόληψη. Τη σπατάλη ε, των ε, τροφίμων και είμαι ικανοποιημένη διότι υπευλήθησαν πολλές τροπολογίες σχεδόν όλες οι ομάδες υπέβαλαν τροπολογίες και για τα απόβλητα των τροφίμων κυρίως, υπευλήθησαν τροπολογίες που θέλουν να ενισχύσουν την ιεράρχηση των αποβλήτων ε, όσον αφορά την πρόληψη πατάλης τροφίμων. Δεν ήταν κάτι που προέβλεπα στην έκθεσή μου, αλλά πιστεύω ότι έπρεπε να το υποστηρίξω. Λοιπόν, όσον αφορά τα, το σπατάλι των τροφίμων, θέλουμε να μειώσουμε ε, να μειώσουμε και τις πατάτες των τροφίμων και τη ρήπανση των ε, θαλασσών. Λοιπόν, ακολουθούμε μια γραμμή η οποία ήδη είχε χνηλατηθεί προηγουμένω. Άλλε τροπολογίε έχουν παρόμοια προσέγγιση για τα βασικά μέσα για την πρόληψη της παραγωγή αποβλήτων και για την ευνόηση τη ε, καινοτομία, τη βιομηχανική παραγωγή και τη καινοτομία. Για την μείωση των αποβλήτων. Στις συνεδρίες των σκιωδών τι επόμενε εβδομάδε θα συζητήσουμε την αυξημένη ευθύνη των παραγωγών. Εδώ έχουν υποβληθεί πάρα πολλές τροπολογίες, καμιά φορά σε σαφή αντίθεση μεταξύ τους και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για σύγκληση απόψεων, έβρεση κοινού παρανομαστού, σε γενική αρχή. Όσον αφορά την αυξημένη ευθύνη των παραγωγών, εξακολουθώ να υποστηρίζω την ανάγκη να υπάρχουν ελάχιστε προδιαγραφέ και απαιτήσει που βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελάχιστε απαιτήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ακολουθήσουμε τη σωστή προσέγγιση. Αυτή είναι η θέση μου. Παρουσιάστηκαν όλες οι απόψεις και αντικρουόμενες, άρα πρέπει να βρούμε σύγκληση όσον αφορά την ενίσχυση της αγοράς των ε, πρώτων υλών και των δευτερογενών υλών. Ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η αγορά αυτή. Γνωρίζουμε ότι μόνο ε, τυπικά επίσημα έχουμε πρόταση αναθεωρήσεως της οδηγίας για τα απόβλητα, αλλά η εμβέλεια η πολιτική είναι πολύ πιο φιλόδοξη και όχι μόνο πολιτική φιλοδοξία, θέλουμε να ευνοήσουμε τη μετάβαση προ μια κυκλική οικονομία. Γι' αυτό η αγορά των πρώτων υλών και δευτερογενών υλών είναι στο επίκεντρο. Και το προαπαιτούμενο για μια αγορά αυτών των πρώτων και δευτερογενών υλών είναι ο υποχρεωτικό χαρακτήρα τη του διαχωρισμού των αποβλήτων. Διότι δεν κάνουμε το διαχωρισμό και δεν υποχρεώσουμε τι χώρε να ακολουθήσουν τη διαφοροποιημένη συλλογή των αποβλήτων, τότε θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτές οι αγορές. Από αυτή την πλευρά ε, είμαι πολύ ικανοποιημένη διότι οι ομάδες υποστήριξαν σχεδόν όλες οι ομάδες, σχεδόν όλες μπορώ να πω, υποστήριξαν την πρότασή μου για την πρόληψη της καταργήσεως των ρητρών όπου η συλλογή, η διαφοροποιημένη, η ξεχωριστή των αποβλήτων προβλέπεται μόνο αν τεχνικά και περιβαλλοντικά και οικονομικά είναι κάτι βιώσιμο. Όλοι πιστεύουμε λοιπόν ότι ή μάλλον αυτό το σύστημα ε, που ευνοεί, τις παρε... την παρέκκληση και όλοι γνωρίζουν ότι πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από αυτό. Ενδιαφέρουσες τροπολογίες υπευλήθησαν λαμβάνουν υπόψη τη δυσκολία των αεροκατοικημένων περιοχών. Ήταν ένα σημείο που δεν το είχα περιλάβει, αλλά είναι αρκετά σημαντικό. Και εξίσου σημαντική είναι η επέκταση των υποχρεώσεων συλλογής της διαφοροποιημένης ε, συλλογής των οργανικών αποβλήτων. Και από αυτή την άποψη υπάρχουν πολλές τροπολογίες που ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση. Βασικό θέμα είναι των στόχων για την αύξηση των ποσοτήτων των πρώτων υλών και των δευτερογενών υλών που διατίθεται στην αγορά που διαφορετικά θα πήγαιναν χαμένες. Όσον αφορά τους στόχους, θέλω να είμαι σαφέστατη. Επαναλαμβάνω εν ονόματι εμού προσωπικά και της ομάδας σοσιαλιστών και δημοκρατών ότι υποστηρίζουμε πλήρως το ψήφισμα ποιητικά είναι που ψηφίστηκε πέρσι από το Κοινοβούλιο όπου ζητήσαμε εκεί στόχους σαφείς 70% ανακύκλωση και προετοιμασία νέας χρήσης ανάμεσα μέχρι το 2030 των αστικών αποβλήτων 80% των συσκευασιών και 5% ε, των ε, περιτυλιγμάτων. Λοιπόν, ε, όχι όλες οι ομάδες παρουσίασαν τροπολογίες επ' αυτού, αλλά είμαι ότι η θέση του Κοινοβουλίου δεν αλλάζει από τη μια χρονιά στην άλλη. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που εγκρίναμε και ψηφίσαμε πέρσι είναι κάτι που για μας εξακολουθεί να είναι αφετηρία. Πολλές τροπολογίες υπευλήθησαν για υπο για την προετοιμασία της χρήσεως. Είναι ένα επιχείρημα που δεν είχα λάβει υπόψη. Με έτοιμη να το συζητήσω αυτό, μάλιστα και όδης, όπως και τα ανακύκλωση των βιοποβλήτων και ε, ε, την ανακύκλωση των διαφόρων βιομηχανικών ελαίων. Μετά είναι η μέθοδος υπολογισμού, οι ορισμοί που είναι θέματα προς εξέταση. Επαναλαμβάνω τη σημασία να έχουμε και κοινό ορισμό του αστικού αποβλήτου και πρέπει να έχουμε μοναδική μέθοδο υπολογισμού που φαντασίζεται σε ένα μοναδικό τρόπο, μοναδική μέθοδο υπολογισμού. Παρουσιάστηκε μία πυρία συνδυασμών, άπειρες, άπειροι συνδυασμοί υπευλήθησαν, ε, πέρα και από τα όρια της φαντασίας και θα πρέπει να βρεθεί όμως ένα πλαίσιο, είναι ευαίσθητο σημείο, εγώ θα ήθελα σαν βαθμό μέτρησης να έχουμε ε, το σημείο στο οποίο γίνεται η ε, κατεργασία του αποβλήτου, τελικό στάδιο της ανακύκλωσης. Μια διευκρίνηση. Μιλάμε εδώ, και το ξέρουν οι σκιώδεις και οι άλλοι συνάδελφοι, ότι εδώ συζητάμε για δημοτικά τέλη, αστικά τέλη, περίπου 7-9% του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να κλείσει ο κύκλος πρέπει να περάσει και να περάσουμε σε πραγματική κυκλική οικονομία πρέπει να θεωρήσουμε μηχανικό απόβλητο και το εμπορικό απόβλητο. Είναι η ιδέα που υποστηρίζουν πολλές πολιτικές ομάδες και θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει για το 2018 μία πρόταση για τους στόχους. Αυτά ήταν τα σημεία για τα οποία επιβλήθησαν οι περισσότερες τροπολογίες. Θα ήθελα από τη συζήτηση να κατανοήσω ποιες είναι οι προτεραιότητες των συναδέλφων. Πιστεύω όμως ότι η δουλειά που ξεκινήσαμε είναι επικοδομητική και γι' αυτό πιστεύω ότι θα βρούμε καλή θέση του Κοινοβουλίου και τελικά θα καταφέρουμε να πετύχουμε, να θεσπίσουμε μια καλή νομοθεσία. Ευχαριστώ. Και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε με τους ε, σκιώδεις εισηγητές από τις πολιτικές ομάδες και ξεκινάμε με τον Καλ Χάιντς ε, Φλόρεντς από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την κυρία Μποναφέ είναι εξαιρετικό το έργο το οποίο έχει φέρει σε πέρας. Δεν ξέρω αν είναι να έχουμε 1900 τροπολογίες για ένα τέτοιο θέμα. Εδώ τίθεται ένα θέμα του πώς μπορούμε να, να τα διαχειριστούμε όλα αυτά. Θυμάμαι την έκθεση για το Ρίτς που είχε φτάσει τις ε, χίλιες σελίδες. Ε, εν πάση περιπτώσει, ίσως χρειάζεται να υπάρχει και μία από τη δική μας ε, πλευρά μία αυτοσυγκράτηση. Έρχομαι στην ουσία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα, οι πρώτες υλε οι οποίες ε, χρησιμοποιούνται πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται. Αυτά είναι μια προτεραιότητα και όχι μόνο για εμάς αλλά και για τι επερχόμενες γενναίες. Γιατί η Ευρώπη δεν έχει πλούτο πρώτων υλών και οι χώρες από τις οποίες παίρνει από τις οποίες παίρνει πρώτες η Ευρώπη δεν είναι ιδιαίτερα πολιτικά σταθερές και δεν είναι εξασφαλισμένη η δυνατότητα εφοδιασμού. Έχουμε λοιπόν προβλήματα και πολιτικά και όχι μονάχα το ηθικό καθήκον να αντιμετωπίσουμε σωστά τα, τα απόβλητα της πρώτες που μπορούν να ανακτηθούν. Πολλές χώρες έχουν ακόμα χωματερές οι οποίες δεν μπορούν από τη μια μέρα στην άλλη να καταργηθούν. Αλλά όπως λέει η Κομισιόν πρέπει να σταματήσουν και οι υποστηρίξεις για χωματερές ή για εγκαταστάσεις ε, καύσεως. Αυτό το οποίο νομίζω όμως ότι θα πρέπει να γίνει πιο σαφές στις εκθέσεις αυτές γιατί έχω παρακολουθήσει από πολύ καιρό την πολιτική για τα απόβλητα και ξέρω ότι δεν έχουν εφαρμοστεί πραγματικά οι οδηγίες στην κατεύθυνση αυτή. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι έχουμε κάνει και εμείς. Υπάρχουν οδηγίες οι οποίες εδώ και 22 χρόνια δεν έχουν προχωρήσει και εδώ τίθεται το θέμα πολλές φορές των ορισμών. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι έχουμε πολλές ιδέες που διατυπώνουν οι συνάδελφοι για την αντιμετώπιση των ε, αποβλήτων. Αλλά όσο δεν έχουμε ένα καλό τρόπο, ένα σωστό τρόπο να καταμετρούμε το πώς γίνεται η αξιοποίηση, η ανακύκλωση των αποβλήτων και όσο δεν έχουμε στοιχεία για τα πόσα απόβλητα εξάγονται ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα επακριβώς και ίσως το ποσοστό ανακύκλωσης είναι πολύ μικρότερο από ό,τι πιστεύουμε. Επομένως δεν ξέρω αν αν θα πρέπει να ακολουθήσουμε την Κομισιόν που θέλει να αυξήσει τα ποσοστά ανακύκλωσης ή να ακολουθήσουμε την φιλοσοφία που ακολουθεί η Γερμανία που λέει να αφήσουμε τις, ε, τα ποσοστά αυτά ε, ανακύκλωσης σταθερά. Ε, αυτό πιστεύω ότι ίσως είναι καλύτερο για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις οι οποίες ήδη έχουν χαράξει μια στρατηγική για την ανακύκλωση με οριζόντα το 2025-2030. Η, αυτά που λέει λοιπόν η κυρία Ποναφέν πιστεύω ότι είναι σωστά ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτήν την ε, νοοτροπία η οποία μας οδηγεί στις ε, χωματερές και στην απλή καύση των ε, αποβλήτων. Βλέπουμε τι γίνεται και με τα τρόφιμα παραδείγματος χάρη, τα οποία απορρίπτονται και πιστεύω Νομίζω ότι η ευθύνη του παραγωγού ενός αγαθού για την μελλοντική του ανακύψη πρέπει και αυτή να ληφθεί υπόψη. Όταν κάποιος παράγει ένα πλαστικό υλικό θα πρέπει να έχει κάποια ευθύνη για αυτό το προϊόν. Αλλά όταν έχουμε ένα νέο, παραδείγματος χάρη, πλυντήριο, το οποίο έχει παραχθεί τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν τόσες πολλές ε, ουσίες που είναι μέσα, τόσα πολλά υλικά τα οποία οδηγούν σε ε, σε, τα οποία είναι απαραίτητα για τις λειτουργίες του πλυντηρίου και δεν μπορούν να αντικατασταθούν με τη νέα τεχνολογία, εκεί υπάρχουν δυσκολίες να μπορέσει να ανακυκλωθεί αυτό το πλυντήριο και εκεί δεν έχει πραγματικά νόημα το να πούμε ότι είναι υπεύθυνο για την ανακύκλωση όλων αυτών των προϊόντων, όλων αυτών των υλικών, των συστατικών στοιχείων ο κατασκευαστής. Αυτό είναι ακόμα και επικίνδυνο τελικά. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει και ένα καλύτερο, μια καλύτερη πρόταση ενοδικού χάρτη για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Φυσικά θέλουμε όλοι να υπάρχει αυτή η ανακύκλωση. Για προϊόντα από χάλιβα πραγματικά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Αλλά για πολλά άλλα προϊόντα, για πολλά άλλα συστατικά που είναι συνθετικού χαρακτήρα είναι πολύ πιο δύσκολο το πρόβλημα αυτό. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς συνθετικά προϊόντα στη βιομηχανία μας. Παραγωγή για ένα, για ένα μοτέρ ανεμιστήρα. Χρειάζεται μια ορισμένη ποσότητα καυσίμου παραδείγματος χάρη ένας ε, ανεμιστήρας, ένας ανακυκλωτής αέρα. Αν έχουμε όμως ανακυκλώσιμα υλικά μπορεί αυτό να σημαίνει ότι θα καταναλώνει πολύ περισσότερο καύσιμο. <clears throat> Αν έχουμε χάρη μέταλλο το οποίο είναι βαρύ και όχι πλαστικά συστατικά τα οποία θα είναι πιο ελαφρά. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μια ισορροπία για τα θέματα αυτά και γι' αυτό θα πρέπει να τα κρατήσει υπόψη της όλα αυτά τα θέματα και η συγγήτρια Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι θέλουν να αφήσουν απ' έξω τελείως την δυνατότητα ε, καινοτομίας των επιχειρήσεων με τον επιβάλλουν άκαμπτες ποσοστώσεις και εν πάση περιπτώσει εγώ θέλω να τονίσω ότι είμαι, χαίρομαι για τις εργασίες της εισηγήτριας και ελπίζω θα μπορέσουμε μέσα στις χρονικές ε, προθεσμίες που έχουμε να βρούμε κάποια συμβαστική λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας την εισηγήτρια, την ευχαριστώ θερμά. Τη συγχαίρω, διότι είναι αφοσιωμένη στο έργο της. Προσπαθεί 100% σημαντικότατο θέμα Υπάρχουν πολλές τροπολογίες, ίσως πάρα πολλές, αλλά και εγώ είμαι ενόχος. Και εγώ υπέβαλα ούκο λίγες, αλλά είναι πολύ σημαντικό θέμα για όλους. Οι διαπραγματεύσεις θα είναι μακροχρόνιες, θα έχετε την υποστήριξή μου και αν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να σπαταλούμε είναι χρόνος. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Γι' αυτό λοιπόν ακούγοντας τις φήμες που έρχονται από το Συμβούλιο περί αναβολής του καθορισμού στόχων για τα απόβλητα, αυτό είναι σίγουρα κάτι ανησυχητικό. Νομίζω ότι οι προτάσεις που έχουμε μπροστά μας εξετάστηκαν, έχει μελετηθεί ο αντίκτυπος των προτάσεων, έχουμε ήδη σπαταλήσει αρκετό χρόνο αποσύροντας την πρώτη πρόταση. Αν ξεκινήσουμε τώρα πάλι την υπονόμευση και αυτής της πρότασης, θα είναι πολύ αρνητική εξέλιξη και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να στείλει ένα σαφέστατο μήνυμα. Πρέπει να δείξουμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε, ότι δεν θέλουμε να κολυσιεργήσουμε. Και σε όλες τις πολιτικές ομάδες συμφωνούμε. Χρειάζεται η μετάβαση αυτή προς μια κυκλική οικονομία. Είναι οικονομική ανάγκη αυτή. Εξαρτώμεθα από την εισαγωγή πρώτων υλών, πολύ, οι πρώτες ύλες εξαντλούνται, και με ταχύ ρυθμό. Άρα δεν έχουμε επιλογή, δεν μπορούμε να παραμείνουμε ως έχουμε. Πρέπει να στηρίξουμε την κυκλική οικονομία, να την προωθήσουμε και να μην θέσουμε τροχοπέδι. Όσον αφορά τα απόβλητα και τη διαχείριση αυτών, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτιώσεων. Τον Ιούνιο είχα πει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα. Υποβάλαμε τροπολογίες προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση Δεν μπορούμε να περιμένουμε δώρα τον Άι Βασίλη, είναι νωρίς ακόμα. Έχουμε κατάλογο όμως δώρων ούτως που θα θέλαμε να μας φέρει ο Άγιος Βασίλης. Είχαμε την πρώτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2014. Χρειαζόμαστε περισσότερες φιλοδοξίε, φιλοδοξίες, χρειαζόμαστε μία και μοναδική μέθοδο μέτρηση. Ε, μέτρησης. Τονίζεται η πρόληψη, η διαχωρισμένη ε, συλλογή των αποβλήτων και τα βιολογικά απόβλητα και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τη θαλάσσια ρήπανση μέχρι το 2030 και θέλουμε να επεξεργαστούμε και το θέμα των, των αποβλήτων τροφίμων και ότι θα πρέπει και οι παραγωγοί να συμμορφωθούν με τις προσπάθειες και θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστοι κανόνες που θα ισχύουν για όλους. Χρειαζόμαστε ισότιμες συνθήκες για όλους. Εάν θέσει κανείς φιλόδοξους στόχους, μπορεί να τους πετύχει μόνο με τη συμμετοχή των παραγωγών. Είναι ύψης της σημασίας αυτό. Τώρα οι χωματερές πρέπει να εξαλειφθούν σταδιακά. Δεν νομίζουμε ότι ανακυκλώσιμα απόβλητα πρέπει να καταλήγουν σχωματερές άνευ κατεργασίας και δεν θα πρέπει να υποστηρίξει μια τέτοια πρακτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέποντας οι διάφορες τροπολογίες, όσον αφορά τα προαναφερθέντα σημεία, ε, έχουμε περιθώρια να συμφωνήσουμε. Όσον αφορά τα τελευταία δύο σημεία που ανέφερα, ίσως τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Και γι' αυτό θα σας πω πού βρισκόμαστε για μία ακόμη φορά. Νομίζω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα συμβάλλουν στην προσπάθεια. Και αναφέρομαι στην τροπολογία μου 1016, ε, εκπλήσωμε που βλέπω ότι κανένας άλλος συνάδελφος δεν επέβαλε παρόμοια τροπολογία. Δεν μπορούμε όμως να επιτρέψουμε πρώτες ύλες για άλλα 20 χρόνια να σπαταλιώνται. Βέβαια, μιλάω από τη δική μου εμπειρία, στη δική μου χώρα, αλλά νομίζω ότι έχουμε επαρκή εμπειρία και τεχνογνωσία στις χώρες εκείνε που έχουν μείνει πίσω, να εξασφαλίσουμε ότι αυτέ οι χώρε μπορούν να προλάβουν το επίπεδο, να φτάσουν στο επίπεδο των άλλων χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και θα κάνω ό,τι μπορώ στι διαπραγματεύσει για να πείσω του συναδέλφου. Μετά, έχουμε και έναν συνδυασμένο στόχο, προετοιμασία για εκ νέου χρήση πρώτων υλών, ανακύκλωση από την άλλη, Βλέποντα την οδηγία πλαίσιο όμω, βλέπετε ότι χρησιμοποιήσει και η προετοιμασία για αυτό θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε ένα άρθρο, ανεξάρτητα από το καθεστώς που έχουν. Το ένα που θεωρείται προϊόν και το άλλο απόβλητο και οι δύο δραστηριότητες έχουν κοινό στόχο παρόλα αυτά. Και αυτή είναι η τροπολογία με 958. Και παραπέμπω σε αυτήν την τροπολογία. Και συνδυασμένος στόχος δεν έχει λογική στην οδηγία πλαίσιο ότι γίνεται διάκριση μεταξύ συσκευασίας μιας χρήσης και συσκευασίας περισσότερων χρήσεων. Αν έχεις έναν ενιαίο συνδυασμένο στόχο, θα έχεις αφύσικα υψηλά στοιχεία, αριθμητικά στοιχεία και θα απομακρυνθούμε από το στόχο της ανακύκλωσης. Άρα δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία του να έχουμε ευρωπαϊμένο, ευρωπαϊκό ε, στόχο για το επίπεδο ε, ε, εκ νέου χρήσεως συσκευασιών και αυτή είναι η τροπολογία μου 981. Τώρα κλείνοντα. και εγώ φιλοδοξώ να έχουμε τελικά μια ξεκάθαρη νομοθεσία, όχι πολύ άκαμπτη. Έχω κι εγώ το κίνητρο να κινηθώ προς το στόχο όπω οι συνάδελφοι και θέλω να συνεργαστώ επικοδομητικά με την εισηγήτρια για να καταλήξουν σε ένα κείμενο το οποίο θα το υποστηρίξουν ε, οι περισσότεροι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο και αυτό χρειαζόμαστε για συνομιλίε με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ και τον Μάκερ ο κύριο Στόρβαλς για την Άλντε. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Συνήθως δεν αρχίζω με συγχαρητήρια. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντα της εισηγητρίας η κυρία Μποναφέ και στη διάρκεια των ε, συναντήσεων με τους κοιόδη ηγητές ήταν καλά οργανωμένος και πλήρης γοητείας και αυτό βεβαίως συμβάλλει τα μάλα. Μπορείτε να διαβάσετε και ανάμεσα στις γραμμές των όσων εκφωνώ. Νομίζω ότι καλά λειτουργεί η ομάδα των διαπραγματευτών. Νομίζω ότι κινούμαστε πάνω σε μια καλή τροχιά. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, υπάρχουν διαφορετικές προσωπικότητες, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχουν συζητηθεί τα πράγματα έως τώρα αποτελούν, αποτελεί καλό παράδειγμα του ότι οι θέσεις δεν είναι ιδεολογικά άκαμπτες. Καλά τα πάμε λοιπόν και αν μπορέσει η διαδικασία να παραμείνει ανοιχτή για κάποιο αριθμό μηνών ακόμη, νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα αξιόλογο έγγραφο και καλύτερο από αυτό το οποίο επεξεργάζεται για την ώρα το Συμβούλιο. Έχουμε βέβαια και κάποια γενικότερα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Προβλήματα τα οποία συνήθως αντιμετωπίζουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα πρέπει να αποφασίσουμε δηλαδή σε ποιο επίπεδο θα νομοθετήσουμε. πρόβλημα που σχεδόν πάντα αντιμετωπίζουμε, γιατί είναι διαφορετικές και οι παραδόσεις των χωρών μελών ε, από τη σκοπιά αυτή. Αν μπούμε στην μικροδιαχείριση, για την οποία αναφέρθηκε πριν ο Μάρκ, δηλαδή μικροδιαχείριση, δηλαδή φτιάχνουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ταυτόχρονα ψάχνουμε να βρούμε και που είναι τα κενά ανάμεσα στα κλαδιά του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. Και όπως ακούσατε και από τους άλλους και ηγητές, η στάση μας είναι αισιόδοξη. Και μοιραζόμαστε και τις ευθύνες. Ε, πρέπει όμως να τονίσω και τουλάχιστον ένα πρόβλημα που έχουμε. Η κυρία Μποναφέ αναφέρθηκε στα απορρίμματα τροφίμων. Σοβαρό πρόβλημα αυτό. Βλέπουμε για παράδειγμα στα σούπερ μάρκετ. Αναγκάζονται τα σούπερ μάρκετ να κάνουν μια επιλογή. 5.000 διαφορετικά είδη, 25.000 διαφορετικά είδη. Και στα υψηλής ποιότητας ας πούμε σούπερ μάρκετ έχουν και 25.000 διαφορετικά είδη και οι ποσότητες που τελικώς καταλήγουν στα σκουπίδια τροφίμων είναι πολύ υψηλε, Πολύ μεγάλες. Στη Φιλανδία κάναμε ένα πείραμα. Μειώσαμε τον αριθμό των ειδών που πόλουν τα σούπερ μάρκετ. Και είδαμε να μειώνεται ποσοστιαία ή ποσότητα των ε, απορριμμάτων. Όμως αν πάμε έτσι θα αντιμετωπίσουμε μεγάλη αντίσταση γιατί θα πούμε τότε στους επιχειρηματίες των μεγάλων σούπερ μάρκετ ότι πρέπει να μειώσουν τα είδη που πολλούν στα καταστήματά τους και μπορείτε να φανταστείτε με τι ενθουσιασμό θα υποδεχτούν την, ε, το έτοιμά μας αυτό. Έχουμε λοιπόν διαφορετικές απόψεις και μεταξύ των σκιωδών εισηγητών. Αυτό εξαρτάται και λίγο από το από πού προέρχεται ο καθής. Αρπαχτήκαμε λίγο με τον Μάρκ εχθές σχετικά με το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς πυκνότητα πληθυσμού 400 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ή ένα άτομο ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο που υπάρχει και αυτό σε ορισμένα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ναι, ε, θα μαλώσουμε κιόλα. όμως όπως είπα και στην αρχή έχουμε εμπιστοσύνη στην κυρία Μποναφέ ότι δηλαδή θα τα καταφέρει να κατευθύνει το σκάφος σε ήσυχα ύδατα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ να ξεπεράσω αυτά που είπε ο κύριο Τόλβατς σε σχέση με το έργο της εισηγήτριας. Χάρη σε αυτό η έκθεση έχει ένα υψηλό επίπεδο φιλοδοξίες, γιατί φυσικά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πράγματι χρειάζεται να υπάρξει βοήθεια, να βελτίωση. Υπάρχουν κάποιες ε, τροπολογίες τις οποίες έχουμε καταθέσει για το ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη αντιμετώπιση των αποβλήτων όπως έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε και στο Κοινοβούλιο της χώρας των Βάσκων και κάνουμε και σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα από τα θέματα τα οποία θέλουμε να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα και δεν έχει τονιστεί ιδιαίτερα είναι η αντίθεσή μας στην καύση υλικών τα οποία είναι ανακτήσιμα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει νομοθεσία ώστε να απαγορευτεί αυτή η πρακτική, ώστε να μην δίδονται κονδύλια για εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων. Κάτι ακόμα το οποίο είναι σημαντικό για μένα είναι ότι η διαχείριση των αποβλήτων δεν είναι μονάχα θέμα των κρατών μελών. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν πολλές φορές αρμοδιότητες στον τομέα αυτό και είναι κυρίως αυτές οι οποίες προωθούν προγράμματα καλύτερης διαχείρισης των αποβλήτων. Θέλουμε λοιπόν στι τροπολογίε αυτέ να υπογραμμίσουμε τη σημασία να υπάρχει συνεργασία όλων των επιπέδων διοίκηση και επομένω να υπάρξει ουσιαστική αναγνώριση του ρόλου των τοπικών αρχών που είναι οι πιο κοντινέ στον πολίτη. Επίση, άλλα σημεία τα οποία έχουν οδηγήσει συζήτηση, σε συζήτηση μέχρι στιγμή, τονίζω ότι εμεί θέλουμε να έχουμε μία ενιαία μέθοδο για την κατάρτιση των στατιστικών, εάν πρόκειται να πετύχουμε στόχους οι οποίοι είναι φιλόδοξοι, με στόχο όχι μόνο να υπάρχει εναρμόνιση στη συλλογή και κατάρτιση των στατιστικών, ώστε, αλλά και ώστε κανείς να μην, μπορεί να μαγειρεύει τα στοιχεία και να παρουσιάσει στοιχεία τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Για το σημείο λοιπόν αυτό, όπως και η, για την υποχρέωση της διαλογής των αποβλήτων, Νομίζω ότι αυτή η οδηγία δεν πρέπει να αφήσει κανένα παρατηράκι, καμία δυνατότητα να παρακάμψει κανείς αυτή την οδηγία, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη συστημική αλλαγή, η οποία θα προωθήσει πραγματικά την κυκλική οικονομία. Γι' αυτό μαζί και με άλλους συναδέλφους προσπαθήσαμε να αφαιρέσουμε ορισμένες ε, ε, ρήτρε οι οποίε είναι σε υποθετικό επίπεδο, εάν συμβεί κάτι δηλαδή θα γίνει κάτι άλλο, ώστε να είναι υποχρεωτικά όλα αυτά τα στοιχεία και να μπορούν να γίνονται οι απαραίτητε ενέργειε. Επίση, είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε δεσμευτικού ε, στόχου, όπω είπαν και άλλοι συνάδελφοι, ακόμα και στόχου οι οποίοι είναι μερικού χαρακτήρα για το 2025. Και αυτοί οι μερικοί στόχοι κατά την άποψή μα, είναι σημαντική, ιδίως σε ό,τι αφορά τα τροφιμικά απόβλητα και τα απόβλητα τα οποία ρηπαίνουν τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Θα ήθελα επίσης να πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας εμπλέξει όλους για να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη μας είναι αρμόδια σε ό,τι αφορά την εξαγωγή αποβλήτων να εμποδίσουν αυτή την εξαγωγή. Πρέπει λοιπόν να είναι σαφής ο στόχος ότι θα πρέπει σιγά σιγά να σταματήσουν να υπάρχουν χωματερές όχι απλώς να μειωθούν αλλά να εξαφανιστούν τελείως και η Κομισιόν θα πρέπει να προσθέσει και ένα στόχο σε σχέση με το συνολικό ε, όγκο ε, αποβλήτων που μπορούν να πηγαίνουν σε χωματερές ο οποίος να καταμετράται σε κιλά ανά άτομο. Θα πρέπει λοιπόν να δίνονται και κίνητρα στις χώρες οι οποίες παράγουν μεγάλο όγκο αποβλήτων να τον μειώσουν με αυτόν τον τρόπο. Κάτι ακόμα το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι οι τροπολογίες μας προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι χρειάζεται να υπάρχει και μια προληπτική προσέγγιση. <clears throat> Νομίζω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες έχουν τονίσει ότι πρέπει να προλαμβάνουμε τη δημιουργία αποβλήτων, αλλά φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την προγραμματισμένη παλαίωση, μάλλον την, ε, το να ξεπερνιέται μια τεχνολογία με τρόπο σχεδιασμένο για τα προϊόντα αυτά, ώστε να χρειάζεται να ανανεώνται. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η ευθύνη των κατασκευαστών, ώστε τα, οι πρώτες να μην κατασπαταλούνται με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύουμε λοιπόν και όπως είπε και η κυρία Μποναφέ ότι ο ελάχιστος ε, κοινό παρονομαστή δεν πρέπει να είναι ελάχιστος. Θα πρέπει να είναι ένας φιλόδοξος κοινό παρονομαστή. Ήταν πολύ, πολύ μεγάλο το έργο που έχουμε να φέρουμε σε πέραση οι συγγητέ και οι σκιώδει συγγητές. Έχουμε ένα κείμενο το οποίο έχει πολύ μεγάλε δυνατότητε, Έχουμε μια μεγάλη ε, συνένεση σε πολλά σημεία και εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι φιλόδοξη αυτή η έκθεση. Ξέρω τώρα ότι δεν αρέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τη λέμε ότι πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη, αλλά εμεί έχουμε εντόπιον μα ένα νομοθετικό πακέτο το οποίο μπορεί πράγματι να δώσει τα ενάυσματα για μια κυκλική οικονομία για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τι πρώτε ύλε και τα υλικά με πιο βιώσιμο και ευφυή τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να πω μιλώντας εκ μέρου του Πρασίνου Σκιώδου Συσηγητού να πω στην κυρία Μποναφέ ότι τους την ευχαριστούμε για την έξοχη δουλειά που έκανε. Το κείμενο που έχουμε μπροστά μας πιστεύουμε ότι ακολουθεί πράγματι τη σωστή κατεύθυνση. Δεν θέλω να επαναλάβω τα υποθέντα από τους συναδέλφους σας και ηγητής για τη γνωμοδότηση για το πακέτο στην Επιτροπή Ήτρε θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποια σημαντικά θέματα, τα οποία θεωρούμε από κοινού κρίσιμου σημασία στην Επιτροπή Ήτρε. Πρώτα απ' όλα να τονίσω τη σημασία της συνέπειας μεταξύ των στοιχείων του πακέτου και όσον αφορά τους ορισμούς στόχους και τα κίνητρα Καμιά φορά διάφοροι τομεί συζητούνται σε διαφορετικέ διαδικασίε. Στην Επιτροπή Ήτρε είδαμε ότι χρειάζεται να καταβληθεί προσπάθεια να ακολουθηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Άλλο σημείο. Να διευρυνθεί το πεδίο από τα αποκλειστικά τακιακά απόβλητα και τα δημοτικά απόβλητα και συμπεριλάβουμε και τα βιομηχανικά απόβλητα με συγκεκριμένους επαρκείς στόχους και πιο φιλόδοξο, ε, φιλόδοξους στόχους ε, και για τα απόβλητα και για τα επίπεδα ανακύκλωσης. Πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά εθνικά προγράμματα και μετρήσεις στα κράτη-μέλη. Δεν αρκεί γενικό στόχος. Πρέπει συγκεκριμένα να θέσουμε στόχους για τα κράτη-μέλη. Υπάρχει επίσης ανάγκη για υποχρεωτική συλλογή δύο αποβλήτων. Είναι σημαντικός τομέας. Το είδαμε και από τη συζήτηση. Πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Καλύτερη υποπτία των επιδόσεων των κρατών μελών. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν αρκεί να καθορίζονται στόχοι για τα κρατημέλη και μόνο. Χρειάζεται έγκαιρη προειδοποίηση και σχετικοί μηχανισμοί, συγκεκριμένη δράση σε περίπτωση κινδύνου μη συμμορφώσεως. Πρέπει να εξασφαλίσουμε και κάτι άλλο, ότι διαφοροποιημένη συλλογή ο διαχωρισμός δεν αφορά μόνο τις χωματερές αλλά και από την καύση. Δηλαδή τα απόβλητα που δεν πάνε πλέον στη χωματερή πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν καταλήγουν και στην καύση για να καταλήξουμε στον τελικό απότερο σκοπό της κυκλικής οικονομίας. Χρειάζεται και κατάλογος εργαλείων για τη μετακίνηση προς την κυκλική οικονομία. Στο το πακέτο. Να δώσουμε κίνητρα για τα δευτερογενή, δευτερογενείς πρωτεσίλες και διάφορα υποχρεωτικά σχήματα για τη συμμόρφωση. Θα πρέπει να έχουμε σφαιρική προσέγγιση. Μέσω μέτρων για ιεράρχηση των αποβλήτων. και χρειάζονται και τα σχετικά μέτρα για αυτή την προσέγγιση. Και ο πότερος στόχος της κυκλικής οικονομίας είναι από καύση και χωματερές να κινηθούμε προς ανακύκλωση, εκ νέου χρήση και πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, που είναι και ο τελικός σκοπός του πακέτου που επεξεργαζόμαστε. Ευχαριστώ. Ο κ. Πεντιτσίνη για το EFTD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τη συνάδελφο Μποναφέ. Έκανε πολύ καλή δουλειά. Είναι σαφές ότι ακολουθούμε καλό δρόμο. Συνεργαζόμαστε άριστα οι ε, και σκιώδεις οι Να προσέξουμε το θέμα της πρόληψης. Αναφερόμενος όχι τόσο στο κείμενο που επεξεργαζόμεθα στο Κοινοβούλιο, αλλά σε εκείνο που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θυμάμαι πολύ καλά ότι όταν ετοιμάσαμε την έκθεση πρωτοβουλίας στοχεύσαμε στην εξάλληψη των επιδοτήσεων για το ρηκτά καύσιμα. Είναι θεμελιώδες αυτό για την πρόληψη. Να επενθυμίσω ότι αυτές οι επιδοτήσεις είναι περίπου 5-3 ευρώ το χρόνο είναι περισσότερα από ό,τι χρησιμοποιούνται στον κόσμο για την υγεία. Και αυτό επηρεάζει κατά πολύ την επιτάχυνση και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Δεν μιλάμε μόνο για την ενέργεια, αλλά και για τα δευτερογενή προϊόντα, όπως είναι τα πλαστικά. Όσο υπάρχουν κίνητρα και επιδοτείται ε, αυτή η παραγωγή δημοσία, τα παραδοσιακά πλαστικά πάντα εμπορικά θα είναι σε θετική θέση σε σύγκριση με ένα οικολογικό πλαστικό ή και καινοτόμο πλαστικό. Και τα παραδοσιακά πλαστικά θα μπορούσαν ποτέ να ενταχθούν στην κυκλική οικονομία που θέλουμε. Θέλω να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Επεσεργάστηκε μια πρόταση στο Κοινοβούλιο. Ψήφισε τη θέση του γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το ζήτημα όμως δεν το συμπεριέλαβε στο κείμενο. Τώρα έχει ενταχθεί. Και τουλάχιστον υπάρχει στήριξη των ομάδων. Πάω σε λεπτομέρειες τώρα, συγκεκριμένα σημεία. Ορισμοί. Δεν θα σταθώ πολύ εδώ. Στο τέλος θα πετύχουμε συμβιβασμό. Και χάρη στη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Τώρα ορισμός των αποβλήτων καλώς τα εμπορικά από τα βιομηχανικά απόβλητα να διαχωριστούν. Διότι τώρα είναι σε έναν κοινό ορισμό. Και δύο κατηγορίες δεν μπορούν και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν να είναι δημοτικά απόβλητα στον ορισμό. Ανακύκλωση, ορισμός της ανακύκλωσης, έννοιας ανακύκλωσης. Να δοθεί προσοχή. Να μην μπει μία έννοια πρόθεσης της ανάκτησης ενεργείας μέσω αναεροβικής ζύμωσης. Από τη στιγμή που αυτή η πρακτική δεν εγγυάται την πλήρη ανάκτηση των μετάλλων με τον κίνδυνο εκπομπών μεθανίου που είναι άριο θερμοκηπίου και καμιά φορά εκπέμπεται και διοξείδιο του Δεν θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιείται αυτό. Μετά, καλό θα ήταν να δώσουμε κίνητα σε διαδικασίες που οδηγούν σε ζήμωση αεροβική, οργανική επεξεργασία των αποβλήτων για να καταλήγουμε σε πολτούς ποιότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αλυπάσματα και να μειώσουμε και το, τη χρήση άνθρακος και το βιοκαύσιμα σε μικρές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιείται για γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αναρωβική επεξεργασία διαφοροποιημένων ε, αποβλήτων. Και το μεθάνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τροφοδότηση δικτύων δημοσίων μπορούν μόνο αν είναι αδρανοί να χρησιμοποιούνται σε συσκευασίε τα απόβλητα. Και εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για μονώσεις στα κτίρια. Μετά, όσον αφορά τα απόβλητα των τροφίμων. Η συμβαστική λύση είναι σωστή, σωστή κατεύθυνση. Παρόλο που έχουν διαφωνίες. Αν πρέπει να υπάρχει διασύνδεση με την ιεράρχηση των αποβλήτων. Να επισημάνω μια λεπτομέρεια Έχουμε επιστημονικές μελέτες που δείχνουν οτιδήποτε καλλιέργεια που χρησιμοποιεί ε, έχει 2% ε, άμα δεν ακολουθήσει στη διαδικασία. Οπότε δεν μπορούμε να διατηρήσουμε τη σωστή ιδιότητα των ε, προϊόντων. Δεν γίνεται σωστά η ανακύκλωση. Η αναφορά στην άρχιση των αποβλήτων υιοθετήθηκε και ελπίζουμε να διατηρηθεί και η συμβαστική. Η πρότασή μας θεωρεί ότι μέτρηση πρέπει να έχουμε μέτρησης, ε, σωστές μετρήσεις για τη μείωση της πατάλης και των, ε, της, της παραγωγής ε, των αποβλήτων τροφίμων. Δεν θα, και δεν θα πρέπει επίσης, θα πρέπει να μειώσουμε μέχρι το 2020 να μειωθεί, να μειωθεί η χρήση των χωματερών και των καύσεων. Λοιπόν, στον τομέα των κατασκευών και των οικοδομών πιστεύουμε ότι η αναδιάθρωση, των, η ε, ανακαίνιση των κτηρίων των υπαρχόντων θα πρέπει να ε, προτιμηθεί ε, εν σχέση με την κατεδάφιση και την χρήση των υλικών της κατεδάφισης και για τα νέα κτίρια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλύτερα τα νέα κτίρια να γίνεται λειτουργία σε προσαρμογή με ανακατασκευή αντί να γίνεται κατεδάφιση μα χρειάζεται να γίνεται κάποια διόρθωση. Στο κείμενο πρέπει να απευθύνεται πρόσκληση στα κράτη-μέλη για να συμπεριλάβουν στο κόστος του περιβάλλοντος ένα προϊόν που έχει ε, να λάβετε υπόψη το ίχνος άνθρακα του κάθε προϊόντος και θα πρέπει να υπάρχουν σταδιακές ε, φορολογικά, να δοθούν φορολογικά κίνητρα ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει όσον αφορά τα απόβλητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζάρκ. Κυρία Εισηγήτρια, αγαπητοί συνάδελφοι, η, τε, η αναθεώρηση των τεσσάρων αυτών οδηγιών για τα απόλυτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη μια κυκλική οικονομία. Είναι απαραίτητο να μειωθούν τα απόβλητα. Το να τα χρησιμοποιήσουμε είναι σημαντικό και σαν ενεργειακή πηγή. Όλοι μας θέλουμε να μειώσουμε τα υλικά συσκευασίας που οδηγούν σε απόβλητα. Και σίγουρα όλα αυτά που λέει η κυρία Μποναφέ είναι ορθά σε αυτό το κατεύθυνο. Αλλά παρόλα αυτά οι προτάσεις των τεσσάρων οδηγιών και οι συμβαστικές τοπολογίες έχουν δύο προβλήματα. Καταρχήν υπάρχει μια, μια άρνηση να γίνει η, η τοπικότητα και η επικουρικότητα ο ακρογωνίος λίθος της πολιτικής για τα απόβλητα. Και συγχρόνως υπάρχει το, υπάρχουν τα πλατιά πλοκάμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θέλει να επιβάλλει μια ενιαία στάση σε όλη την Ευρώπη. Αυτό οδηγεί σε προβλήματα παραβίασης σε επικουρικότητας αλλά και σε πρακτικά επίπεδα. Τα εμπορικά και τα δημοτικά απόβλητα δεν είναι τόσο σημαντικά όσο το χαρτί που πετιέται κάθε μέρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεωρείται ότι είναι δημοτικό απόβλητο, ενώ είναι εμπορικό απόβλητο αυτό που πετάνε παραγωγικά τα καταστήματα. Τα θέματα αυτά λοιπόν πρέπει να είναι ζητήματα των κρατών μελών αποκλειστικά. Τα φορολογικά ε, ωφέλη, τα ωφέληματα τα οποία προτείνονται για να είναι κίνητρα για τα κράτη να αντιμετωπίσουν τα απόβλητα παραβιάζουν την αρχή της ε, επικουρικότητας. Οι οδηγίες αυτές λοιπόν θα έχουν ένα μεγάλο βάρος πάνω στους οικονομικούς φορείς χωρίς να αποφέρουν τους απαραίτητους καρπούς. Η καύση δεν ανανεώνει, καταστρέφει. Οι εγκαταστάσεις καύσης της τελευταίας γενιάς επιτρέπουν και την παραγωγή ενέργειας και δεν αφήνουν παρά ελάχιστη τέφρα. Επομένως, δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθούν πλήρως, δεδομένου ότι η χρήση τους και η παραγωγή ενέργειας μπορεί να συγκεντρωθεί καλύτερα σε τοπικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, υπογραμμίζοντας την τοπική αντιμετώπιση και την επίλυση των προβλημάτων σε κάθε περιοχή και όχι γενικά, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια ε, καλύτερη αντιμετώπιση των αποβλήτων και όχι μια κοινή αγορά αποβλήτων όπως θέλει η έκθεση. Ευχαριστώ. Η Σας ευχαριστώ και εγώ θέλω να συνταχθώ μαζί με τους συναδέλφους μου για να συγχαρώ την εισηγήτρια για το πακέτο αυτό της κυκλικής οικονομίας, αλλά θα ήθελα να κάνω και μερικά σχόλια. Λόγω του, της εμβέλειας του θέματος αυτού που μας απασχολεί, δεν πρέπει να συγχαίουμε την ταχύτητα με την βεβαιασμένη ενέργεια σε σχέση με τη δράση που πρέπει να κάνουμε για τα τροφιμικά απόβλητα θα πρέπει να υπάρχει ένας ορισμός ο οποίος καλύπτει όλους από τον αρχικό παραγωγή, παραγωγό ως τους καταναλωτές. Αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα για πάρα πολλά από τα κράτη-μέλη μας. Συγχρόνως όμως θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στην ανάγκη στο να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ απολειών στην παραγωγή και κατασπατάλησης πρώτων υλών. Για μένα δεν είναι σαφής οι ορισμοί και αυτό δεν μας βοηθάει να δημιουργήσουμε μια ιεραρχία για τα απόβλητα και δεν μας βοηθάει να έχουμε και την καλύτερη πρόληψη. Και έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την χρήση τροφιμικών προϊόντων για ανθρώπους που χρησιμοποιείται μετά για διατροφή ζώων και επίσης έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε στην, ε, να δημιουργήσουμε μπορούμε να περάσουμε στην κομποστοποίηση ορισμένων από αυτά τα απόβλητα ή να παραγάγουμε και, και μεθάνιο από αυτά. Επίσης, για την κατάργηση των εγκαταστάσεων καύσης. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση θα οδηγήσει σε μια απλοποίηση των διαδικασιών, απλώς θα οδηγήσει σε προβλήματα ερμηνείας στα κράτη-μέλη η διατύπωση η οποία υπάρχει και εν πάση περιπτώσει δεν θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ξέρουν προς τα που θα πρέπει να κινηθούν στο μέλλον. Τρίτο σημείο, το τέλος της ζωής των αποβλήτων. Και εκεί πάλι αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ένα αποτέλεσμα και να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να έχουμε σαφείς ορισμούς, ενιαίους ορισμούς οι οποίοι δεν επιδέχονται πολλές ε, ερμηνείες διαφορετικές στα κράτη-μέλη και που θα πρέπει να την χάνουν αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των κρατών για τις μεθόδους υπολογισμού και εδώ είμαστε όλοι σχεδόν που έχουμε ζητήσει να υπάρχει ε, ένας υπολογισμός για τον όγκο των αποβλήτων μετά από την πρώτη διαλογή. Αυτό έχει το πλεονέκτημα της, απλότητα της απλότητος και της εφαρμοσιμότητας και μπορεί να βοηθήσει να απλοποιήσει και να κάνει πιο αποτελεσματική την διαδικασία και με τον τρόπο αυτό μειώνουμε και το κόστος γιατί η διαλογή των αποβλήτων στα κράτη-μέλη γίνεται με διαφορετικό τρόπο και διαφορετική οργάνωση. Και τελευταίο θέμα, θέλω να αναφερθώ στον ορισμό του αποβλήτου. Είναι σημαντικό να μιλήσουμε για δημοτικά απόβλητα, αντίθετα με αυτά που είπε ο προηγούμενος ομιλητής, όταν μιλάμε για παρόμοια απόβλητα θα πρέπει να έχουν και σε ποσότητα και σε σύνθεση συγκρίσιμο χαρακτήρα. Αυτό είναι σημαντικό όταν θέτουμε το θέμα της ευθύνης των τοπικών ε, κοινωνιών και φορέων. Δεν πρέπει λοιπόν να ε, ευνοείται η δημιουργία μεγάλων μαζών ε, αποβλήτων γιατί δεν είναι προσαρμοσμένε σε αυτά οι εγκαταστάσει. Ευχαριστώ, λέω Η Κολίν Λάγκεν. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρώτα θέλω και εγώ να ενώσω τη φωνή μου στην έκφραση συγχαρητηρίων προς την κυρία Μποναφέ. Ούτε άλλωστε θα ήθελα τώρα να επαναλάβω όλα όσα λέχθηκαν ήδη. Επισημαίνω ότι για μένα ιδιαίτερη σημασία στην πρόταση έχει και έχω κάνει και σχετικές τροπολογίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενες πρώτες ύλες. Γι' αυτό και πρέπει να αναπτύξουμε μια πολιτική προϊόντων που να λαμβάνει υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις σε όλο τον κύκλο ζωής από την παραγωγή μέχρι και την τελική διάθεση των προϊόντων. Σε αυτή την κυκλική οικονομία οι πρώτες ύλες μετά από το πέρας του κύκλου ζωής να επανέρχονται στον κύκλο παραγωγής. Βεβαίως και ενίσχυση της αποφυγής παραγωγής απορριμμάτων, διότι αυτό θα εξυπηρετήσει και την αηφορία αλλά και θα επηρεάσει και την συμπεριφορά των καταναλωτών. Το σύστημα της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού είναι σημαντικό επίσης στοιχείο. Χαίρομαι λοιπόν για την εισαγωγή των ελάχιστων αυτών απαιτήσεων, διότι είναι σημαντικό να μην αναμειχθούμε εκεί στην κυριαρχία ρυθμίσεως των χωρών μελών. υπερβολικά λεπτομερείς ρυθμίσεις νομίζω ότι θα περιορίσουν με τρόπο αδικαιολόγητο την ρυθμιστική κυριαρχία των, κρατών μελών. Πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη η αρχή της επικουρικότητας. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι εθνικέ ιδιαιτερότητε, χωρί ταυτόχρονα να τεθούν σε κίνδυνο οι ενιαίοι ευρωπαϊκοί στόχοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ο Σκαπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω προφανώς να ευχαριστήσω τη Σιμώνα για την συνεχή της δουλειά, τις άκρες προσπάθειές της. Ε, είναι περίπλοκη δουλειά πάνω από 2.000 τροπολογίες να σε επεξεργαστεί κανείς δεν είναι κάτι απλό. Θα ήθελα να αποφύγω να επαναλάβω τα υποθέντα του συναδέλφους. Θέλω όμως να τονίσω κάποιες πτυχές. Το θέμα των στόχων. Επ' αυτού συμφωνώ απολύτως με τη φιλόδοξη πρόταση της Σιμώνα. Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα σαφές αδιαμφισβήτητο ότι θα περάσουμε οριστικά από την οικονομία τη γραμμική προς μια κυκλική. Είμαι υπέρ και της προτάσεως της ε, αυξήσεως των κυρώσεων των μη συμμορφούμενων κρατών μελών με, με τους στόχους. Όσον αφορά την ευθύνη των παραγωγών, είμαι ανάμεσα σε αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να είμαστε πιο φιλοδόξοι όσον αφορά την ευθύνη. Παρουσίασα διάφορες τροπολογίες από αυτού. Πρέπει να έχουμε ελάχιστα επίπεδα, ελάχιστα διαγραφές ευθύνης. Και ήδη η παραγωγή θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθούν από τις ποινές που συνεπάγεται η μη συμμόρφωση με αυτούς τους ε, στόχους. πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ε, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για σχεδιασμό και χρήση των υλικών και χρήση και σχεδιασμό των προϊόντων προς αυτή την κατεύθυνση από πλευρά παραγωγών. Έτσι θα μειώσουμε στο ελάχιστο, απαραίτητο ελάχιστο την καύση και τις ε, χωματερές, όπως αναφέρθηκε. Πρέπει να επιμείνουμε για μια καλύτερη υποπτία και καλύτερο συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέποντας τα αποτελέσματα τα πενιχρά των εθνικών προγραμμάτων προλήψεως. Κατά την άποψή μου δεν μπορούμε να υποθέτουμε ότι το fact-checking να γίνεται μόνο στο τέλος της διάρκειας του προγράμματος προλήψεως χωρίς να προβλέπεται και ένας έλεγχος και αναθεώρηση ενδιάμεση ε, όσον αφορά τη, τα υιοθετηθέντα μέτρα. Άλλο σημείο που θεωρώ σημαντικό να σταθώ. Η οδηγία για τις συσκευασίες να χρησιμοποιούνται ε, που χρησιμοποιούνται περισσότερο βιολογικά, βιοδιασπόμενα υλικά, αλλά χρειάζεται καλύτερη διείσδυση τεχνολογία στην αγορά για να βελτιωθεί έτσι η λειτουργία του συστήματος της ετικετοθεσίας ε, των βιοδιασπομένων συσκευασιών. Κάτι άλλο. Το food waste, η σπατάλη τροφίμων και των αποβλήτων τροφίμων, υπέβαλε σχετικά πολλές τροπολογίες. Βλέποντας την αύξηση της φτώχειας και την ηθική υποχρέωση που έχουμε όλα να αποφύγουμε τη σπατάλη των τροφίμων. Που τα τρόφιμα είναι απαραίτητα για εκείνους που έχουν, πάσχουν από ένδια. Χρειάζεται εκστρατεία ευαισθητοποιήσεω στα κράτη-μέλη. Πρέπει να δοθούν και φορολογικά και οικονομικά κίνητρα πέραν αυτών για τη συλλογή των ε, προϊόντων που δεν χρησιμοποιούνται στο λιανεμπόριο και στο catering για να μπορούν τελικά να ε, μοιράζονται από ε, φιλανθρωπικούς φορείς. Η κυκλική οικονομία χαρακτηρίζει αυτή τη θητεία. Είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα πρέπει να μας κάνει να διακριθούμε. Μπορούμε να ξανασχεδιάσουμε πραγματικά την κοινωνική διάδροση, να βρούμε ένα νέο τρόπο ζωής. Εύχομαι καλή τύχη στη Σιμώνα για την κυκλική οικονομία ε, και καλή δύναμη για να συνεχίσεις αυτή την περίπλοκη δουλειά που κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε με τους ευρωβουλευτές. Θέλουμε να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μας πει ποια είναι η θέση της για τις τροπολογίες. Και των όσων υπόθηκαν σήμερα στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την Σιμώνα Μποναφέη. Έκανε, κάνει σκληρή δουλειά και την περιμένει ακόμα πολύ σκληρή δουλειά. Ευχαριστώ και τους Ευρωβουλευτές για τον εντυπωσιακό αριθμό τροπολογιών πιστεύω ότι καταδεικνύουν ότι δίνουν προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό. Διαβάσαμε όλες τις τροπολογίες, είτε το πιστεύετε είτε όχι. Και χαιρόμεθα που υπάρχει γενική υποστήριξη για μια φιλόδοξη προσέγγιση, προς μια νέα πολιτική για τα αποβλητά. Η προτεραιότητά μας είναι η ταχεία πρόοδος όσον αφορά τις προτάσεις. Θέλουμε να μας δώσουν τάχιστα αποτελέσματα. Η σημασία της ταχείας εγκρίσεως αναφέρθηκε στην επιστολή του Προέδρου Γιούνκερ και του κυρίου Τίμερμαν στην Επιτρόπου, απευθυνόμενη επιστολή προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, του κυρίου Σούλτς. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εισηγήτρια και τους κοιόδης εισηγητές στην προσπάθεια για συμβιβασμούς, ούτως ώστε γρήγορα να καταλήξουμε στην επιθυμητή συμφωνία όχι μόνο εντό του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά μια συμφωνία θέλουμε γρήγορα και με το Συμβούλιο. Για τους στόχους. Είναι κρίσιμη η σημασία τους για συμφωνία. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να συνδυάσουμε ρεαλισμό και φιλοδοξία και όπου χρειάζεται και δικαιολογείται και να δώσουμε κάποιο χρόνο παραπάνω σε κάποια κάτι μέλη ούτως ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν και αυτά στην προσπάθεια. Ταυτόχρονα σφίγγουμε τα λουριά. Με τον ορισμό για τα δημοτικά απόβλητα θα καλύψουμε περισσότερα απόβλητα. Και με τους στόχους και τους κανόνες περιπολογισμών στοχεύουμε στην εξασφάλιση της μετρήσεως αυτού που πράγματι μπορεί να ανακυκλωθεί όλα τα κρατη Με τις αλλαγές αυτές και τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία ήδη έχουν υψηλό ποσοστό ανακυκλώσεως θα πρέπει να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθεια στην επίτευξη των στόχων που έχουμε προτείνει. Γι' αυτό λέμε ότι είναι φιλόδοξη η πρόταση, αλλά είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων. Όσον αφορά τις ε, παρατάσεις ή ε, τις χρονικές, οι τροπολογίες δεν αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού, έχοντας σαν στόχο το 2020. Ταυτόχρονα, κάποιες τροπολογίες ίσως περιπλέξουν το σύστημα, ίσως μειώσουν την ασφάλεια δικαίου και ίσως αυξήσουν διοικητικό άχθος άνευ σημαντικών θετικών αποτελεσμάτων σε αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, κυρίως των χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα. πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποια κράτη-μέλη χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να συμμορφωθούν. Δεν μπορούμε να μειώσουμε το χρόνο. Εάν καταβάλει προσπάθειες και δεν μπορεί να πετύχει ενδιάμεσους στόχους, να πετύχει μετά πιο υψηλούς στόχους. Επιδεινούται η κατάσταση. Θέλουμε να δώσουμε χρόνο στα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με το χρονοδιάγραμμα. Και αν δεν τα καταφέρουν, έχουμε και άλλα μέσα εάν δεν συμμορφωθούν καλή την πίστη, έχουμε και διαδικασίες κατά παράβαση. Θέλουμε όσον αφορά την εποπτεία ε, να βλέπουμε τι πραγματικά να κυκλούται. Είναι απαραίτητο λοιπόν να μπορέσουμε να κάνουμε την ε, συλλογή Δεν έχει όμω ιδιαίτερο νόημα. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει στη μονάδα ανακύκλωσή, Ίσως να υπάρχουν όμως και ανάμεικτα απόβλητα εκεί, μεικτά απόβλητα και να αντιμετωπίσει καμία δυσκολία. Αν μετρήσει κάνει τι μετρήσεις, κάποιο μπορεί να βρει κατά πόσο η διαλογή γίνεται σωστή. Αν έχουμε σωστή μέτρηση μπορούμε να εντοπίσουμε όλα τα στάδια τη ανακύκλωση να λειτουργούν σωστά. Σε ό,τι αφορά του νέου στόχου που προτείνονται δηλαδή αποφυγή παραγωγής ε, απορριμμάτων, το, ε, ε, μείωση της παραγωγής απορριμμάτων τροφίμων και το καθεσής. Σωστή είναι η στόχη, βεβαίως, και πρέπει αυτά να γίνουν αντικείμενο μελέτης επιπτώσεων και βεβαίως και να συνοδευτούν με μέτρα επίτευξής τους. Εμείς είμαστε υπέρ του να παραμείνει η στόχευση πάνω σε αυτούς τους στόχου που έχουν προταθεί εξ, εξ αρχής και οι νέοι να έχουν και ρεαλιστικές προθεσμίες. Μια και υπάρχει και ρήτρα αναθεώρηση το 2024. Αν θέλετε νέους στόχους, χρειαζόμαστε καλής ποιότητας δεδομένα και καλής ποιότητας μεθοδολογία. Για παράδειγμα, για τα απορρίμματα τροφίμων, αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι είναι σημαντικό να γίνει. Αλλά δεν έχουμε όμως την κατάλληλη μεθοδολογία ούτε τα καλής ποιότητας δεδομένα. Γι' αυτό προτείνουμε να η αναλυθεί δράση για να αναπτυχθεί η σχετική μεθοδολογία και όταν θα την έχουμε πλέον ας επανέλθουμε σε λίγα χρόνια. Δεν είμαι βέβαιος ότι το να μπει ένα στόχος τώρα σε ένα νομοθετικό κείμενο είναι καλή, καλή ιδέα. Το ίδιο για την δημιουργία νέων ορισμών για ιδιαίτερα είδη απορριμμάτων, γιατί μπορεί να έχει σημαντικέ νομικέ συνέπειε. Οι ορισμοί εξυπηρετούν την θέση στόχων και αυτά πρέπει να συμβαδίζουν. Σημειώνουμε με ενδιαφέρον τις διατάξεις σχετικά με, το, με την ε, ε, αυστηρότερη διατύπωση των ε, απαιτήσεων για, τις, για την αποκομιδή πρέπει να γίνεται ξεχωριστά. Από εκεί πρέπει να αρχίζει κιόλας η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων και με τον φθηνότερο δυνατό τρόπο να προσφέρονται και ε, δευτερεύουσες πρώτες ύλες στην βιομηχανία. Ταυτόχρονα θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να είναι τόσο αυστηρές και λεπτομερείς οι ρυθμίσεις που τελικώς να μην είναι βέβαια η έκβασή τους. Ορισμένες από τις εξαιρέσεις θα πρέπει να επιτρέπονται. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία στην διάκριση των απορριμμάτων είναι η αποτελεσματικότητα του συστήματος. Εγώ δεν έχω ε, ενδείξεις ότι υπάρχει κατάχρηση των εξαιρεσεών. Έχετε εσείς ενδείξεις να μας τις θέσετε υπόψη. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να καταστήσουμε βέβαιον ότι τα συστήματα διακρίσεως των απορριμμάτων είναι ξεκάθαρα, απλά για τους πολίτες και ότι πραγματικά ξεχωρίζουν τα απορρίμματά τους. Κάποια ευκαμψία χρειάζεται και στην επιλογή των οικονομικών μηχανισμών. Είναι χρήσιμα κάποια εργαλεία πολιτικής, αλλά ας αποφύγουμε τις σύνταγες. Το είπατε και εσείς. Οι χώρες μέλη μπορεί να μην έχουν διάθεση να εφαρμόσουν όλα, όλους τους ενδεχόμενους μηχανισμούς, αλλά ίσως προτιμούν να ψάξουν να βρουν το σωστό μείγμα των διαφόρων νομοθετικών ε, ρυθμίσεων κλπ. Α υπάρχει ο κατάλογο, αλλά μην επιβάλλουμε στις χώρες μέλη να τα εφαρμόσουν όλα αυτά ταυτόχρονα. Είδαμε και εμεί τι πολλέ ε, τροπολογίε και για την διεύρυνση της ευθύνη του παραγωγού. Συμφωνούμε με αυτά, με τον στόχο αυτό και νομίζω ότι και το Συμβούλιο κινείται προ την ίδια κατεύθυνση. Ας αναζητήσουμε λοιπόν εδώ κάποιες ορθές λύσεις και το γεγονός ότι πολλοί εξημών τονίσατε την ανάγκη διεύρυνση της ευθύνης του παραγωγού με καθιστά αισιόδοξο. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα μέσα για να επιτύχουμε να κλείσει ο κύκλος της οικονομίας. Ας φροντίσουμε να υπάρχει λοιπόν και ισότιμος ανταγωνισμός για όλα αυτά. Υπάρχουν και τροπολογίες που αναφέρονται σε θέματα που είναι πολύ σημαντικά για την κυκλική οικονομία και το πεδίο εφαρμογή βέβαια, για παράδειγμα, απώλειες τροφίμων που ξεφεύγουν όμως από το πεδίο εφαρμογή της παρούσης οδηγίας που έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τα απορρίμματα, ενώ αυτά τα food losses αναφέρονται μάλλον στην αλυσίδα παραγωγής και προμήθειας τροφίμων. Μπορεί μάλιστα να έχουν και το αντίθετο αποτέλεσμα εν τέλει οι τροπολογίες αυτές για την κυκλική οικονομία. Ε, διατάξεις όπως επισήμανση κλπ. Ε, σε ένα νομοθέτημα δηλαδή το οποίο ασχολείται με τα απορρίμματα μπορεί, επειδή τα πράγματα αυτά είναι πολύ περίπλοκα, μπορεί να ε, υποστηβλάβει τελικώς. Χρειάζεται ξεχωριστή ρύθμιση, αυτό θέλω να πω. Και το τελευταίο, και αυτό μας ανησυχεί πολύ, είναι ο αριθμός νέων καθηκόντων και νέων προθεσμιών που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ έχω μετρήσει 10 και μέχρι το 2018 τουλάχιστον μέχρι το 2018-10 και επανέρχονται και έρχονται και άλλες. Θα επανέλθω σε αυτό που είπατε ορισμένοι εξημών για την εφαρμογή. Στα επόμενα χρόνια αυτό που με ενδιαφέρει είναι να επιτύχει η εφαρμογή. Διότι αν χρειαστεί να κατανολώνουμε τον χρόνο μας συντάσσοντας νέα έγγραφα, νέους στόχους, νέες νομικές προτάσεις, νομίζω ότι τελικώς θα χάσουμε στο πεδίο εκείνο της εφαρμογής που ίσως είναι πιο βαρετό αλλά εγώ δεν βλέπω να γίνεται πρόοδος χωρίς επιτυχία στην εφαρμογή ναι. και εκεί πρέπει να διαθέσουμε προσπάθεια και πόρους. Συνολικά, ωστόσο, οφείλω να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένο από το φιλόδοξο πνεύμα που βλέπω να διέπει τη σκέψη σας και αν όντως συμβαίνει αυτό, Νομίζω ότι εν τέλει θα επιτεύχουμε μια ορθή συμφωνία και για τους λόγους αυτούς ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια και απευθύνω έκκληση προς όλες και όλους σας να συνεχίσετε με τρόπον ώστε να επιτύχουμε συμφωνία το δυνατόν συντομότερο. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now we can... Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση δίνοντας το λόγο στην εισηγήτρια για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Κύριε Μποναφέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους που ήταν πολύτιμη και αυτή τη φορά. Επικοδομητικές συνεισφορές, ακριβείς, τεκμηριωμένες και εγώ και οι σκιώδη σίγουρα θα τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Μπορώ να πω ότι υπάρχουν δύο λόγια περισσότερα από άλλα αναφέρθηκαν εδώ. Το ένα ήταν η λέξη φιλοδοξία και η άλλη ήταν η λέξη ευθύνη. Η λέξη φιλοδοξία που τη σημερίστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό με ικανοποιεί. Η πρόταση που υπευλήθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την άποψή μου είναι μια καλή αφετηρία. Αφετηρία που σίγουρα περιέχει στοιχεία τα οποία εμείς ενισχύουμε Εκείνο που διαφάνει είναι ότι όλοι έχουμε πραγματικά τη βούληση για βελτίωση της προτάσεως και να καταλήξουμε στις διαπραγματεύσεις με μια θέση ε, όσο πιο κοινή γίνεται. Φιλοδοξία. Ε, ακούσαμε και τα σχόλια των συναδέλφων ότι δεν σημαίνει να μην είναι κανείς ρεαλιστής. Αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, διότι όλοι οι στόχοι που θέτουμε είναι στόχοι που κατά κάποιο τρόπο παραμένουν ήδη ευέλτιστη πρακτική που εφαρμόζεται σήμερα. Αυτό το λέω για να σας πω ότι η φιλοδοξία μπορεί να είναι ρεαλιστική και θέλουμε η φιλοδοξία της τελικής πρότασης να είναι ρεαλιστική. Η άλλη λέξη που θεωρώ ότι αναφέρθηκε περισσότερο από τις άλλες ήταν ευθύνη. Και εδώ υπάρχουν πολλά σημεία που μας βρίσκουν να συμφωνούμε από αυτά που ακούσαμε κιόλας όσον αφορά τις υποχρεώσεις ε, ε αυτής διαφοροποιημένης συλλογή των αποβλήτων είναι κοινή για την πρόληψη, όλοι συμφωνούμε, ε, έχει σημασία η πρόληψη για τα μέτρα της ενισχύσεως της προλήψεως, για την πρόληψη που θα είναι ένα πρώτο θεμελιώδες βήμα όσον αφορά την ιεραρχία των αποβλήτων, συμφωνούμε όλοι. Και σήμερα ε, επαναλάβαμε τη σημασία που έχει να βασιστούμε επί του food waste όχι μόνο σαν πρόβλημα περιβαλλοντικό αλλά και αδοντολογικό, σπατάλη τροφίμων και τα τροφιμικά απόβλητα. Ε, υπάρχουν κάποια σημεία που διαφάνησαν σαφώς επί των οποίων υπάρχουν αποκλήσεις απόψεων και όπως θα ήταν σωστό και δίκαιο να υπάρχει. Ε, και το, το είπα και εγώ και στην εισαγωγή μου. Οι τροπολογίες έδειξαν ότι υπάρχουν διαφορές ε, είδαμε ότι διαφοροποιούμε στα εξισχέσεις που εκφράστηκαν. Πρέπει να καταλάβουμε προσπάθειες για να καταλάβουμε τι θέλουμε. Μέθοδος υπολογισμού. Και αυτό θέλει επεξεργασία, όχι τόσο όσον αφορά την αναρμόνιση της μεθόδου υπολογισμού που θεωρώ ότι είναι μία από τις έννοιες που θα μπορούσαμε να στηρίξουμε όλοι μαζί όσον αφορά την εισαγωγή των στοιχείων για την προσμέτρηση και του υπολογισμού. Και εκεί μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω προσπάθειε για τον ορισμό του αστικού αποβλήτου. Θέλω να πω ότι ξεκινάμε, ε, υποθέτω σήμερα δεν υπάρχει ορισμό του αστικού αποβλήτου. Και εδώ θα πρέπει να αρχίσει η συζήτηση και από αυτού θα πρέπει να μπούμε στην ε, ουσία και να κάνουμε αξιολογήσει και να συζητήσουμε και τι είναι τα εμπορικά απόβλητα και τα βιομηχανικά απόβλητα. Θα τα ξεργαστούμε όλα αυτά. Πέρα από αυτά τα σημεία που εν μέρη συμφωνούμε, εν μέρη διαφωνούμε, αναφέρθηκε και η λέξη ευθύνη και όχι τυχαία. Επανειλημμένα ακούστηκε η λέξη ευθύνη και δεν είναι τυχαίο αυτό. πιστεύω ότι διεφάνει ότι όλοι αισθανόμαστε την ευθύνη που υπάρχει. Ευθύνη να έχουμε στα χέρια μας ένα σημαντικό εργαλείο για να επαναπροωθήσουμε την περιβαλλοντική πολιτική και τη βιομηχανική της Ευρώπης μας. Και ο παράγων χρόνος όπως υπογράμμισε κάποιος δεν είναι δευτερευούσης σημασίας ο παράγοντας χρόνος δεν είναι μεταβλητή ανεξάρτητη. Αντίθετα, ο παράγον χρόνος είναι ένας παράγον ο οποίος καλεί όλους να καταβάλουν, ε, να αναλάβουν και άλλες ευθύνες μάλλον. Ε, ξέρετε πόσο ε, έχουμε επεξεργαστεί αυτή την πρόταση, όλοι ξέρετε πόσο αναμένεται αυτή η πρόταση και όσον αφορά τη δουλειά που κάναμε, πώς οι ίδιοι εμπλεκόμενοι φορείς εν γέννη όχι μόνο οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις αλλά και τα συνδικάτα, οι ενώσει των βιομηχάνων, των επιχειρηματιών κλπ. Οι ίδιοι πολίτε, όλοι οι φορείς, τα θεσμικά όργανα. Πραγματικά ε, υπήρξε τοποθέτηση ούτω ώστε να υπαρεξετάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τι απόψει των εμπλεκομένων φορέων. Όσον αφορά τους χρόνους, θα πρέπει να προχωρήσουμε με μεγάλη αποφασιστικότητα. Φτάνω και στις επικρίσεις που ακούστηκαν και τις κριτικές που ακούστηκαν. Υπάρχει συμφωνία για την ευαισθητοποίηση του καταναλωτού. Όσον αφορά δηλαδή δημόσιες σχέσεις και η ευαισθητοποίηση μπορεί να οδηγήσει στο να καταλάβει ο καταναλωτής που πρέπει να αγοράζει προϊόντα ανακυκλώσιμα, βιώσιμα προϊόντα. Ε, συμφωνώ με αυτό. Και συμφωνώ όσον αφορά το food waste, επί της αρχής συμφωνούμε όλοι, αλλά αληθεύει ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στην όλη αλυσίδα του food waste. Και χρειάζεται αυστηρότητα όσον αφορά την επεξεργασία των διαφόρων targets. Πρέπει να πω λοιπόν ότι ε, για την άλλη ιδέα ότι δεν λάβαμε υπόψη την επικουρικότητα ακούστηκε αυτή η επίκριση. Θα ήθελα να πω ότι αν η επικουρικότητα είναι αυτή που οδηγεί κάποιε χώρε σήμερα το 90% των αποβλήτων να τα βάζουν στις χωματερέ με σοβαρέ ζημίε για το περιβάλλον και με την απώλεια σημαντικών πρώτων υλών που είναι σημαντικέ για τη χώρα και για την οικονομία τη, ναι, δεν λάβαμε υπόψη αυτή την επικουρικότητα. Αν αντίθετα η επικουρικότητα είναι αυτή που αποφασίζει μια νομοθεσία που είναι σαφής που λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία που υπάρχει στα κράτη-μέλη και τη διαφορά του κράτου μέλου. Και ίσω με επενδύσει και προσεκτικέ πολιτικέ βοηθούνται οι χώρε να πετύχουν του καθοριστέ στόχου, τότε κατά άποψή μου είναι ευφυή χρήση και ευφυή ερμηνεία τη επικουρικότητα. Υπάρχει μια άλλη επίκριση που, με την οποία συμφωνώ, δηλαδή ότι αυτή η τοποθέτηση δεν παράγει οικονομικά ωφέλη. Ίσως δεν κατάλαβα, ίσως να μην κατάλαβα καλά Λοιπόν, επαναλαμβάνω, όπως υπενθύμησε κάποιος συνάδελφος, ότι εμείς εξαρτώμεθα από την εισαγωγή πρώτων υλών και υπάρχουν δύο τρόποι για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε μια παγκοσμιοποιημένη επιθετική αγορά. Πρώτα απ' όλο είναι να συγκρατήσουμε το κόστο ε, εργασία και να το χαμηλώσουμε. Αυτή δεν είναι η ιστορία μα. Άλλο τρόπο να το πετύχουμε αυτό είναι αντίθετα να μειώσουμε το κόστο των πρώτων υλών. Να βασιστούμε στην καινοτομία, στην τεχνολογία που είναι πράγματα στα οποία τα πηγαίνει καλά η Ευρώπη. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι δεν είναι ότι δεν οδηγεί σε οικονομικά ωφέλη αυτό το πακέτο πέρα από την προστινέμενη αξία για το περιβάλλον δημιουργούνται και συνθήκες για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, ένα μοντέλο ανάπτυξης που οδηγεί ευημερία και ποιότητα. Λοιπόν, είμαστε στα μισά του, στα μισά του έργου, της προσπαθίας. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα. Πιστεύω ότι και σκιώδες συζητητές ε, το γνωρίζουν αυτό. Θα πρέπει να προχωρήσουμε, όμως ε, πιστεύω ότι το κλίμα είναι σωστό για να καταλήξουμε σε καλούς συμβιβασμούς. Ε, το αποτέλεσμα της εργασίας εξαρτάται από όλους, Πιστεύω πραγματικά ότι όλοι κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και εντός ε, των χρονικών ορίων που είναι αρκετά περιορισμένα. Τι να πω, πρέπει να ευχηθούμε ότι και το Συμβούλιο θα μας δει σαν παράδειγμα και θα ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή την ταχεία για να καταλήξει το ταχύτερο δυνατό στην έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν την εισηγήτρια για το τόσο σημαντικό έργο που έχει φέρει σε πέρας και νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε εδώ τη συνεδρίασή μας ε, σήμερα. Ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά τους και για τη συμμετοχή τους.